Good afternoon. Καλησπέρα σας και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στην επόμενη ε, συνάντηση, η οποία είναι μια δημόσια κρόση μεταξύ της ΑΦΕΤ και της ε, ΔΡΟΑ σχετικά με την παγκόσμια πολιτική δέσμευση για την ευθύνη ε, προστασίας. Όπως γνωρίζετε, η ευθύνη προστασίας είναι μια παγκόσμια πολιτική δέσμευση, η οποία υποστηρίχθηκε από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ ε, στη σύνοδο, στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του 2005 για την αποτροπή της γενοκτονίας εγκλημάτων πολέμου, εθνοκαθάρσης ε, και εγκλήματα κατά της, ανθ, ανθρωπότητας. Η συγκεκριμένη ακρόαση είναι πολύ έγκυρη δεδομένη της κατάστασης ε, στη Συρία αλλά και σε άλλες χώρες. Κάθε χρόνο λοιπόν η Επιτροπή ΑΦΕΤ ετοιμάζει μια πρόταση για μια σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο ε, για ε, να θέσει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την προετοιμασία για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο συνάδελφός μας από τη Βουλγαρία, Άντρεϊ Κόβατσεφ, ε, ετοίμασε μία έκθεση η οποία εγκρίθηκε στις 30 Μαΐου του ΙΣΑΦΕΤ και μία παράγραφος αναφέρεται στο ζήτημα ευθύνης προστασίας. Η έκθεση λοιπόν καλεί να ενισχύσουμε το ρόλο ε, της ευθύνης προστασίας ως μια σημαντική αρχή ε, στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. να εργαστούμε πάνω στην επίλυση ε, διαμαχών, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη, για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ΟΗΕ για να παίξει το ρόλο του στη βοήθεια προς τις χώρες για την εφαρμογή της ευθύνης προστασίας, αλλά και να προωθήσουμε μια, έναν ευρύ ορισμό ε, για το ε, για την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας και την αρχή της ευθύνης προστασίας. Ε, και ε, τώρα θα ήθελα να δώσω το ε, λόγο στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία. Ο κύριος Παντσέρη δεν μπορούσε να έρθει εδώ και για αυτό το λόγο θα διαβαστούν κάποια σχόλιά του. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι οι δύο επιτροπές μας συνεδριάζουν από κοινού σε αυτή τη δημόσια κρόαση διότι ο Κόφι Ανάν είχε πει ότι ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του σήμερα είναι η πόλεμη του αύριο, του αύριο και ε, νομίζω ότι αυτή η έννοια ευθύνη προστασία είναι πολύ σημαντική για να ε, υπολογίσουμε αν οι κυβερνήσει ε, και οι διεθνεί κοινότητε έχουν κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν στην συνέχεια να προβούν στην στρατιωτική παρέμβαση. Είναι καλό λοιπόν που το συζητούμε αυτό και από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Επιτροπή ε, χαιρόμαστε λοιπόν ε, για το γεγονός ότι έχουμε ανάμεσά μας τον κύριο ε, Σιμόνοβιτς ε, ο οποίος είναι ειδικό σύμβουλος για το ζήτημα ευθύνης προστασίας στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης ε, μία ε, έκθεση για ε, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και της χειρονοκτονίας που θα ψηφιστεί σύντομα και εδώ αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η έννοια της ευθύνης προστασίας. Ήθελα να προσθέσω ότι ε, στο ε, ψήφισμα μας ε, θα πρέπει το, όπου θα συζητήσουμε για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου θα ε, συμπεριλάβουμε και το ζήτημα της ευθύνης προστασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για εμάς. Ε, ο ε, κύριος Σιμόνοβιτς είναι ανάμεσά μας. Θα ακούσουμε αρχικά από αυτόν και στη συνέχεια έχουμε τον καθηγητή Σίμον Άνταμς ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Παγκοσμίου Κέντρου για την ευθύνη Προστασίας από τη Νέα Υόρκη και έχουμε και τον ε, Eric David, ο οποίος είναι από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελών ε, και έχουμε τον κύριο Λέφλερ, ε, ο οποίος που θα μας μιλήσει για το ζήτημα ευθύνης προστασίας. Έχουμε λοιπόν αρκετούς σημαντικούς ομιλητές. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε από εσάς κύριε Σιμόνοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Συμπρόεδρη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους οργανωτές που έδωσαν το θέμα αυτό της ευθύνη της προστασίας στην ατζέντα του σημερινής, σημερινής Σας ευχαριστώ επίσης που με προσκαλέσατε να συμμετάσχω. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να σας, για μένα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις υπάρχουσες προκλήσεις στο θέμα αυτό και να εκφράσω και τις ανησυχίες μου αλλά και τις ελπίδες μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα ο κύριος Σάιμον Άνταμς είναι συνάδελφος και φίλος συνεργάζομαι συχνά στην Ιγάρ και χαίρομαι που είναι εδώ μαζί μας ε, χαίρομαι επίσης που είναι εδώ ο εξαιρετικός ακαδημαϊκός ο κύριος Νταβίδ ε, η σύνθεση αυτή δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη να εργαστούμε και από το θέμα της ε, ευθύνη για προστασία. Οι διεθνείς οργανώσεις, οι ενώσεις, η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνικές οργανώσεις, οι ε, ακαδημαϊκοί, αλλά και τα κράτη-μέλη. Το επίπεδο κατανόησης ό,τι αφορά το R2P, την ε, ευθύνη για την προστασία ε, ποικίλια από ό,τι ξέρουμε μεταξύ των ευρωβουλευτών. Θα κάνω λοιπόν μια μικρή εισαγωγή και μετά θα εξηγήσω και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Το 2005 το αποτέλεσμα ε, μιας παγκόσμιας διάσκεψης ήταν ένα έγγραφο ε, ένα έγγραφο το οποίο προσπέραψαν αρχηγοί 100 κυβερνήσεων και που αναφέρει την αρχή της ευθύνης προστασίας. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι μια υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους να προστατεύει πληθυσμού στο έδαφος του από ειδεχθεί εγκλήματα, από γενοκτονίες, από εγκλήματα πολέμου, από εγκλήματα κάτω της ανθρωπότητας και από εθνοκαθάρσεις. Εάν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να παράσχει αυτή την προστασία μόνο του, τότε έχουν την υποχρέωση τα λοιπά κράτη-μέλη να παράσχουν συνδρομή για να μπορέσει να γίνει, να χώρα αυτή η προστασία. Αν ένα κράτος μέλος αποτύχει στο να προστατεύσει τον πληθυσμό στο εδαφός του ή εφόσον το ίδιο το κράτος εμπλέκεται σε αυτά τα εγκλήματα, τότε υπάρχει συλλογική ευθύνη όλων των κρατών Έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τους πληθυσμούς και να το κάνουν αυτό μέσω των Ηνωμένων Εθνών ε, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια δράση που μπορεί να πάρει πολλέ μορφέ. Ειρηνικά μέτρα, διαμεσολάβηση, αλλά και ε, κυρώσεις ε, και βεβαίως ως ίστατη ε, λύση ή ένοπλη επέμβαση. Αυτή εξ αρχή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει ότι θέλει να προστατεύσει, να προσπίσει αυτήν τη δέσμευση. Αναφέρεται άλλωστε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2013. Ίσως ε, το πιο ισχυρό ψήφισμα για την ε, ευθύνη προστασίας που έχει ποτέ εγκριθεί από οποιοδήποτε διακυβερνητικό όργανο. Βεβαίως ε, το σχέδιο δράσης το οποίο ζητούσε το ψήφισμα που με το όνομα συνένεσης, κονσένσους για, το, για την ευθύνη προστασίας δεν τελεσφόρησε ποτέ, αλλά ε, είχαμε πολλές δράσεις μετά από αυτό το ψήφισμα. Ο κύριος Λεύλε ήταν, έγινε το εστιακό σημείο, το σημείο εστίαση, σημείο επαφής ε, για τα ζητήματα ευθύνη προστασία, ενίσχυση συστημάτων έγκαιρη περιοδοποίηση ε, τις εξωτερικέ εξωτερικές υπηρεσίες υπό το ακρονίμιο PRISM και επίσης ε, η στρατηγική για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης ε, που αναφέρεται στην ε, ευθύνη προστασίας και πρόσφατα επίσης είχαμε συνένεση γύρω από τα ζητήματα ανάπτυξης όπου και εκεί ε, γίνεται αναφορά στην ευθύνη προστασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη, διότι η ευθύνη προστασίας αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή σημαντικές προκλήσεις. Αντιμετωπίζουμε μια αλλαγή, μια μετάβαση από μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται σε αξίες και στο διεθνέ δίκαιο ε, σε μια πολιτική που βασίζεται μόνο σε εθνικά συμφέροντα. Η αποδυνάμωση της παγκόσμιας αλληλεγγύης και του πολυμερούς χαρακτήρα ε, αποτυπώνεται και στο θέμα της ευθύνης προστασίας. Η ευρωπαϊκή υποστήριξη στην ευθύνη προστασίας ε, εκτιμάται ιδιαίτερα από τα Ηνωμένα Έθνη. αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ε, θεωρώ ότι η ευθύνη προστασίας βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Γιατί? Διότι υπάρχει μια σοβαρή ε, απόκληση ανάμεσα ε, στις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και τις τάσεις ιδεχθών εγκλημάτων. Η ευθύνη προστασίας έχει επαναληφθεί πολλές φορές η αρχή αυτή, πάνω από 100 ε, προσώπους στα ε, Ηνωμένα Έθνη, στην Γενική Συνέλευση, επαναλαμβάνουν τη δεσμευσή τους γύρω από αυτή την αρχή. Πάνω από 50 ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρουν στην ευθύνη προστασία, πάνω από 20 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, σχεδόν η κάθε ειρνευτική αποστολή περιλαμβάνουν στην εντολή τους την προστασία των πολιτών. Όμως στην πράξη, στην πραγματικότητα έχουμε αύξηση ε, στις φρικαλαιότητες. Έχουμε αύξηση στις σειράξεις, έχουμε αύξηση της απώλειες πολιτών και, τα μεγέθη έχουν αυξάνει. Τα μεγέθη των, του αριθμού των, του άμαχου που πεθαίνει ε, στις σειράξεις. Είτε ε, αυτό γίνεται ως παράπλευρη απώλεια, είτε επειδή ε, είναι άμεσος στόχος. Είναι εγκλήματα αυτά, είναι εγκλήματα πολέμου και όταν έχουμε συστηματική χρήση αυτών των πρακτικών, τότε μιλάμε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ε, οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε όλους μας. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, 21 εκατομμύρια, και ένας μεγάλος αριθμός αυτών ε, ψάχνουν ε, ένα ασφαλή λιμένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν είτε να εφαρμοστεί πραγματικά αυτή η αρχή είτε να χάσει το νόημά της. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Παρότι ε, οι τάσεις είναι αρνητικές, υπάρχει ένα momentum αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια συγκυρία που μπορεί να μας επιτρέψει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση, να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Καταρχήν έχουμε νέο γενικό γραμματέα στην Ηνωμένα Έθνη που έχει δώσει έμφαση στην πρόληψη. Η ευθύνη προστασίας αποτελεί μέρος της συνολική ατζέντα πρόληψης και υπογραμμίζεται η σημασία της πρόληψης των ε, εγκλημάτων και των φρικαλαιοτήτων. Εάν οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει και αφορούν την προστασία και την πρόληψη ε, τελεσφορήσουν, τότε μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση των προσπαθειών για την πρόληψη και θα έρθουν πιο κοντά οι τρεις πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών. Ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά θα έρθουν πιο κοντά, πιο κοντά στα πλαίσια της πρόληψης των ε, εγκλημάτων πολέμου. Εγώ έχω λάβει μια εντολή, έχω αυτή τη θητεία εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο και προέρχομαι από μια άλλη θητεία όπου μου βοηθό του Γενικού Γραμματέα για τα Στήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα, μια επιχειρησιακή θέση. Ε, επισκέφθηκα σχεδόν όλους ε, τις χώρες όπου λαμβάνουν χώρα ε, οι δεχθεί εγκλήματα και έμαθα ότι ο αριθμός των εκθέσεων ή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ δεν είναι αυτό που μας δείχνει ε, το βαθμό επιτυχίας μας. Ε, το βαθμό επιτυχίας κρίνεται από το τι γίνεται επί τόπου. Αυτή είναι η εμπειρία που έχω από την προηγούμενη θητεία μου και την φέρνω μαζί μου αυτή την εμπειρία, τη φέρω μαζί μου εδώ, σε αυτή τη νέα θητεία η ευθύνη προστασίας λοιπόν πρέπει να πάρει μια πρακτική μορφή. Για να εφαρμοστεί η ευθύνη προστασίας χρειάζεται λογοδοσία για το θέμα της πρόληψης. Να σας πω και ένα καλό νέο. Ο Γενικός Γραμματέας δέχτηκε ως θεματική στα πλαίσια της έκθεσης ε, για την ευθύνη προστασίας το θέμα της λογοδοσίας. Αυτό είναι μία ε, αλλαγή, έτσι. Περνάμε δηλαδή από μια αλλαγη ετσι περναμε δηλαδη συζήτηση σε μια πιο επιχειρησιακή φάση σε ό,τι αφορά την, την αρχή της ε, ευθύνης προστασίας. Ε, χθες υπέβαλα την έκθεση με τίτλο «Εφαρμογή της ευθύνης προστασίας, λογοδοσία για την πρόληψη, στο Γενικό Γραμματέα. Θα το εξετάσει, στη συνέχεια θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των Εθνών και στις 6 Σεπτεμβρίου στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενική Συνέλευση, θα έχουμε μια συζήτηση διαδραστική ε, γύρω από αυτή την έκθεση. Βεβαίως, η έκθεση αυτή δεν έχει ακόμα πάρει το πράσινο φως, αλλά μπορώ να σας πω ήδη από τώρα τις κεντρικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, προς τις διακυβερνητικούς φορείς και τις δεσμεύσεις κλειδιά του γραμματέα, της γραμματείας των ΗΠΑ και του ίδιου του Γενικού Γραμματέα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Υπάρχει το θέμα της ευθύνης προστασίας και των σχετικών σημείων εστίασης θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με την πρόληψη ε, φρικαλαιοτήτων. Επίσης, ε, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να περιλαμβάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου για την πιθανότητα φρικαλαιοτήτων ε, εγκλημάτων στις περιοδικές εκθέσεις προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες μηχανισμού και εδώ βεβαίως ε, κρίσιμοι μηχανισμοί είναι οι συζητήσει στα κοινοβούλια παραδείγματος χάρη ε, έτσι ώστε να γίνει αξιολόγηση κινδύνου αλλά και να συζητηθούν τα μέτρα πώς δηλαδή μπορεί, να, να μειωθούν τα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πρόληψη φρικαλαιοτήτων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει συζήτηση και τον προπολογισμό. Κατά πόσο δηλαδή δίδονται επαρκή χρήματα για την πρόληψη. Ε, μπορεί να γίνει στα πλαίσια εκθέσεων ε, για τι ε, ενώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή μέσω κάποιων δημοσιογραφητών, μπορεί να γίνουν και θεματικέ συζητήσει, ένα κοινοβούλιο για την πρόληψη Φρικαλαιοτήτων ή να οριστεί κάποια επιτροπή, υποεπιτροπή, ad hoc, που θα εστιάζει ε, αποκλειστικά στο θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες συστάσεις πρέπει να σας πω ότι είχα ήδη ε, επαφή με κάποια δίκτυα, δίκτυα βουλευτών, ομπουτσμαν, ε, διαμεσολαβητών, καθώς και Ινστιτούτα και, και θεσμούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι έτοιμοι όλοι αυτοί να πιέσουν για την πρακτική εφαρμογή αυτών των συστάσεων και στο καθένα από αυτά τα δίκτυα ε, θα δώσω κάποια στοιχεία πολύ πρακτικά για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές τις συστάσεις. Και τώρα θα περάσω στους διακυβερνητικούς μηχανισμούς. Γενική Συνέλευση υιοθέτησε διαδικαστικό ψηφισμό ώστε να τοποθετηθεί η ευθύνη προστασίας ε, καθώς και για την πρόληψη φρικτών ε, εγκλημάτων στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό θα μετατρέψει την ε, άτυπη συζήτηση σε μια επίσημη συζήτηση περί ευθύνης για προστασία και για πρόληψη φρικαλωτήτων και ε, σίγουρα αυτό θα δώσει μεγαλύτερο κύρος ε, στη συζήτηση όπως επίσης ε, το ίδιο εφέ θα έχουν και τα πρακτικά αυτής της επίσημης συζήτησης. Το να τοποθετηθεί αυτή η περιοδική αναθεώρηση μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόληψη των φρικαλαιοτήτων, το να χρησιμοποιούνται εκθέσεις για να καταγράφεται εκτίμηση κινδύνου, ε, καθώς και τα μέτρα που χρειάζονται. Το ίδιο το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ε, στη διάρκεια συζήτησης ε, των εκθέσεων αυτών, καθώς και στις συστάσεις που θα περιλαμβάνονται εκεί. Ο στόχο δεν είναι να ε, δακτυλοδείξουμε τα κάτι μέλη όπου, μπορεί να υπάρχουν κενά όσον αφορά την πρόληψη ε, φρικαλωτήτων, αλλά να κινητοποιήσουμε ενέργεια και στήριξη και στήριξη και κρατών μελών ε, ώστε να καλύψουν αυτά τα κενά. Να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ε, ανοιχτή συζήτηση για το ρόλο πρόληψης των ε, φρικαλαιοτήτων, ε, μία, τουλάχιστον μία ανοιχτή συζήτηση για το Συμβουλίο Ασφαλείας για αυτό το θέμα και να δίνεται και μία έμφαση στην λογοδοσία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στα υπόλοιπα κράτη-μέλη όσον αφορά τη δράση και την μη και την αδράνεια για την πρόληψη των φρικαλαιοτήτων. Και τώρα να πω κάτι για τη γραμματεία και για τις δεσμεύσεις του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει ένα, ε, μια αξιολόγηση όσον αφορά τις επιδόσεις μας ε, στη, όσον αφορά την ευθύνη προστασίας. Να προσφέρει δε ε, στοιχεία για το τι διαθετικά μέτρα λαμβάνονται ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για τέτοιου είδους κλίματα, να βελτιώνει τη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες, τα διάφορα τμήματα του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνα για την πρόληψη των εγκλημάτων, αλλά και να δεσμευτεί, δεσμευτεί και να χρησιμοποιήσει το άρθρο 99 του χάρτη, ώστε οι κίνδυνοι ε, ε, φρικών εγκλημάτων να συζητώνται και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Για να ολοκληρώσω. Ξέρω ότι με κύριοι Ευρωβουλευτές έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε ε, σε αυτές τις συστάσεις και όσον αφορά γενικότερα την ευθύνη προστασίας. Και αυτό διότι είστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είστε και βουλευτές. Σε αυτές τις, ε, δύσκολου δύσκολους καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, παγκόσμιο ρόλο στην υποστήριξη της ευθύνη προστασίας, αλλά καθώς και στην λογοδοσία για την πρόληψη των ε, εγκλημάτων. Οι βουλευτές έχουν να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά τη λογοδοσία και πέρα από ένα μακρύ ε, ε, ε, κατάλογο μέτρων που εσείς οι ίδιοι έχετε συμπεριλάβει στο κοινοβουλευτικό ψήφισμα του 2013 για την ευθύνη για προστασία, ίσως θα μπορούσατε να σκεφτείτε και κάποια επιπλέον μέτρα, ίσως να θέλετε να καθιερώσετε μια ετήσια συζήτηση για την πρόληψη φρικαλαιοτήτων και για το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, ακόμα και να χρησιμοποιήσετε ήδη υφιστάμενα βήματα που βρίσκονται στην ημερησία σας διάταξη για την εκτίμηση των κινδύνων και για την αξιολόγηση των μέτρων που μπορούν να αναλυφθούν ε, κοιτάζοντας προς τα μέσα, προς τις ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή της Ένωσης αλλά και προς τα έξω στις γειτονικές σας χώρες αλλά και στον ε, κόσμο ολόκληρο. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πάνω-πάνω στον κατάλογο των περιοχών όπου ίσως συμβούν ε, ε, φρικτά εγκλήματα. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι καμία χώρα δεν είναι απολύτως απαλλαγμένη από τέτοιου είδους κινδύνους. Ίσως λοιπόν η Επιτροπή αλλά και η Υποεπιτροπή που συμμετέχετε εδώ αλλά και άλλες επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου ε, θα μπορούσαν να συζητήσουν το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Τέλος. Όταν ένας ευρωβουλευτής μιλάει, ο κόσμος τον ακούει Γι' αυτό σας καλώ να χρησιμοποιήσετε το κύριο σας και την απήχησή σας εντός των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και εθνικά και διεθνώς ώστε να ενισχύσετε την ευθύνη προστασίας. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, προσδοκώ την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Είστε και συμπατριώτες. Είμαι πολύ περήφανη για τα όσα είπατε ε, και ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις στη διάρκεια της συζήτησης. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ερικ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Έχετε το λόγο και έχετε 15 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές αυτής της συνεδρίασης που με προσκάλεσαν. Σκοπεύω να σας κάνω μια παρουσίαση που όπως ε, θα φαντάζεστε είναι κάπως ε, ακαδημαϊκού τύπου. Λυπούμε ευθύνη προστασίας όσον, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Ε, θα, η ομιλία μου περιλαμβάνει δύο τμήματα. Ένα πρώτο τμήμα που αποδεικνύει ότι είναι μια παλαιά υποχρέωση, η ευθύνη προστασίας, η υποχρέωση προστασίας είναι κάτι πολύ παλιό και από την άλλη πλευρά θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες οι νομικές που απορρέουν από αυτήν την υποχρέωση. Καταρχάς είναι παλιά αυτή η υποχρέωση η οποία ε, ανήκει στο κράτος. Ε, μπορούμε ας πούμε, να ανατρέξουμε στην ε, κήρυξη ανεξαρτησίας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών όπου σε εκείνη τη διακήρυξη σε ένα απόσπασμα λέει ότι η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις μάλλον, ε, δημιουργούνται από τους ανθρώπους για να εγγυώνται το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και της αναζήτηση της ευτυχίας. Αυτό ήδη λοιπόν το 1776 Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άρθρο 1 λέει ότι στόχο των Ηνωμένων Εθνών είναι και στην παράγραφο 3 λέει συγκεκριμένα και παραθέτω να υλοποιήσει τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους. Εδώ έχετε άλλη μια πηγή που όπως βλέπετε δεν είναι διόλου πρόσφατη. Για να δούμε αυτό το χρονολόγιο, φτάνουμε στην ε, Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το στο 16ο εκτιμώντα του προημείου λέει ότι τα κρατημέλη έχουν δεσμευθεί να εξασφαλίζουν έχουν δεσμευθεί να εξασφαλίζουν σε συνεργασία με τον ΟΗΕ τον καθολικό και πραγματικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά Ήδη υπάρχουν, έχουμε εδώ δηλαδή τις βάσεις του κανόνα αυτού και αν όχι τον ίδιο τον κανόνα. Έχουμε το σύμφωνο που αφορά τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα ε, του 1966 που λέει ότι τα κράτη που ανήκουν σε αυτό το σύμφωνο ε, δεσμεύονται να σέβονται και να εγγυώνται σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στην επικράτειά τους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το σύμφωνο αυτό και η Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θεσπίζεται από αυτό το σύμφωνο σε μια γενική παρατήρηση που υιοθετήθηκε το 2004, λέει ότι αυτή η νομική υποχρέωση σεβασμού και εγγύησης όλων των δικαιωμάτων σημαίνει για, όλους τους, ε, για όλα τα κράτη υποχρέωση ταυτόχρονα αρνητική, δηλαδή να μην ε, θίξουν αυτά τα δικαιώματα και μια, και μια θετική υποχρέωση, δηλαδή την λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε αυτά τα δικαιώματα να μην ε, είναι ψευδιστήσεις ή δικαιώματα, φαντάσματα. Και έπειτα έχουμε ένα καθεστώς ε, σε μια διατύπωση νομικού τύπου που πολύ γνωστή και από τους διεθνιστές. Έχουμε και την ε, δέουσα επιμέλεια, due diligence, πολύ γνωστός όρος, 1870 ήδη υπήρχε αυτός ο όρος ε, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές είναι οι πηγές, οι παλές πηγές αυτής της υποχρέωσης. Πρόσφατες πηγές Έχουμε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το 2004 όσον αφορά την κατάσταση στο Νταρφούρ, όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας θυμίζει και παραθέτω πως ε, Καταρχάς, η Σουδανική κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει τους πληθυσμούς που βρίσκονται στην επικράτειά της, να σέβεται τα ανθρωπίνα δικαιώματα και να διατηρεί την δημόσια τάξη. Και κυρίως το τελικό κείμενο του παγκο... της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του 2005 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως στην παράγραφο 138 επισήμως λέει αυτό το που λέγεται responsibility to protect, ευθύνη προστασίας, ε, ευθύνη κάθε κράτο είναι να προστατεύει από τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ευθύνε, που συνίστανται στην πρόληψη, πρόληψη αυτών των εγκλημάτων συμπεριλαμβανόμενη της πρόληψης μέσω της ε, λήψης των απαραίτητων και κατάλληλων μέτρων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υιοθετήσει και παραθέσει αυτούς τους κανόνες πάνω από 60 φορές έκτοτε, είτε για γενικά θέματα όπως η προστασία των αμάχων και των παιδιών, ε, κατά τη διάρκεια νόμπλα σειράξεων, λέμε ότι καταρχάς η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να, ε, να λαμβάνει την ευθύνη αυτή τη προστασία όσον αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατία, ή την πρόληψη των συγκρούσεων ή την διακίνηση όπλων μικρού ή ε, επίσης το έχει επαναλάβει με την ευκαιρία διαφόρων άλλων ε, ε, περιπτώσεων, ταραχών, Κονγκό, Γινέα Μπισάου, Λιβύη, Ακτή Ελεφαντοστού, Γεμένη, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Μαλή, Βοσνία Ζεκοβίνη, Συρία, Σουδάν, Δαρφούρ, Νότιο Σουδάν, Λιβυρία, σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις έχουμε ξανά και ξανά, λες και είναι κάποιο, ε, κάποια λιτανία, ένα είδος πιστεύω, αυτή την υπενθύμηση στις κυβερνήσεις ότι βασικά δικός τους ρόλος είναι να εξασφαλίσουν την προστασία των πληθυσμών που βρίσκονται στην επικρατειά τους και δεν ανήκει αυτό μόνο στα κράτη αλλά και στη διεθνή κοινότητα η διεθνής κοινότητα, που είναι μια, ένας όρος πολύ γενικός και αόριστος, αλλά βασικά σημαίνει το σύνολο των κρατών τα οποία λαμβάνονται υπόψη ως ένας θεσμός. Και πάνε, επανέρχομαι στο 2005 και την ε, διάσκεψη κορυφής της Γενικής Συνέλευσης, όπου λέει και παραθέτω η διεθνής κοινότητα επίσης οφείλει στο πλαίσιο του ΟΗΕ να χρησιμοποιήσει τα διπλωματικά, ανθρωπιστικά και άλλα ειρηνικά μέσα ε, σύμφωνα με το άρθρο 6 και 8 του χάρτη ε, με στόχο να προστατευθούν οι πληθυσμοί από γενοκτονία, κλίματα πολέμου κτλ. Και μετά προστίθεται μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας σύμφωνα με το χάρτη και το κεφάλαιο 7 από εκεί προχωρά ακόμα πιο μακριά και γίνεται δηλαδή έτσι μνήα στην υιοθέτηση από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας αναγκαστικών μέτρων ώστε να υλοποιηθεί, να δεθεί σε εφαρμογή αυτή η προστασία. Και τώρα αυτή η υποχρέωση ε, ε, μεταφράζεται και σε πράξη μέσω κάποιων εκθέσεων όπως αυτή για τη Ρουάντα το 1999, η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη σφαγή της Εμπρένιτσα επίσης το 1999 και την έκθεση της αποστολής υψηλού επίπεδου στον Ταρφούρ το 2007 όπου κάθε φορά γίνεται ακούραστη υπενθύμηση αυτής της υποχρέωσης προστασίας. Ο κανόνας είναι σαφής, δεν νομίζω πως εδώ έχω φεύρει τον τροχό, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες που παράγουν νομικά από αυτό τον κανόνα είναι ένας κανόνα διεθνού δικαίου. Υποχρέωση προστασία, υποχρέωση που βαραίνει τα κράτη-μέλη και τα διεθνεί θεσμού να εξασφαλίζουν την προστασία των πληθυσμών έναντι των φρικτών εγκλημάτων που μπορεί να διαπραχθούν. Αυτός είναι ένας κανόνα διεθνού δικαίου και ο μη σεβασμός αυτού του κανόνα επιφέρει ευθύνη των κρατών ή των ε, ε, ε, λοιπόν διεθνών οργανισμών. Και εδώ αναφέρομαι στο σχέδιο έκθεση τη Επιτροπή Διεθνού Δικαίου σε αυτό το τομέα ότι είναι κάτι το θεωρητικό. Ε, αλλά κάποιες φορές περνάμε και στην πράξη. Αλλά για την ώρα δεν έχω δίποτε κάμια υπόθεση η οποία να έχει πάει σε κάποιο διεθνές δικαστήριο όπου θα αμφισβητηθεί η ευθύνη ενός κράτους ή της διεθνούς κοινότητας επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Και εγώ βεβαίως προσωπικά προσπάθησα να πείσω το, τη Ρουάντα να επιτεθεί εναντίον του ΟΙΕ ενώπιον της Επιτροπής ε, Καταγγελιών που είχε προβλεφθεί ε, στην συμφωνία που, που, που συνήφθη ανάμεσα στη Ρουάντα και τον ΟΗΕ όταν δηλαδή η αποστολή του ΟΙΕ κατέφτασε στη Ρουάντα για να εξασφαλίσει μεταξύ άλλων την προστασία των αμάχων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κιγκαλή, και υπήρξε μια ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στην κυβέρνηση της Ρουάντα και του Γενικού Γραμματέα του ΟΙΕ που αμέσως απέρριψε αυτή την προσφορά πολύ θαραλέα θα έλεγα λέγοντας ότι ναι όλα αυτά είναι θέματα διεθνούς δικαίου και η Επιτροπή Καταγγελιών δεν έχει αρμοδιότητα γι' αυτό. Ήταν κάπως παράξενο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΑ να επιβεβαιώνει πως η Επιτροπή αυτή δεν ήταν αρμόδια. Νομίζω πως δεν ήταν δική του δουλειά να το πει, η ίδια η Επιτροπή θα έπρεπε να το πει αυτό γιατί έχει την <laughs> αρμοδιότητα της αρμοδιότητας όπως λέμε μεταξύ νομικών. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να έχει πολύ σημαντικέ νομικέ επιπτώσεις, δηλαδή την αμφισβήτηση των κρατών ή των οργανισμών που δεν ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά του, Και τελευταία υπάρχουν ενδιαφέρουσε. Ε, ε, συζητήσεις ε, γιατί τα κράτη έχουν μεν αυτή την υποχρέωση προστασίας. Είναι λίγο κενή ο νοήματος αυτή η διατύπωση, αλλά θα προστίθεται ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση προστασίας. Και έτσι, σε σχέση με ένα ψήφισμα που αφορά την ΑΕΤ, στις, ε, λέει για τις αστυνομικές δυνάμεις δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουν στη διαθεσία τους τις απαραίτητες ε, ε, τα, τα απαραίτητα κονδύλια για να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές προστασίας. Ε, και το ίδιο για τη Σομαλία. Πιο πρόσφατα το Συμβούλιο Ασφαλείας χρησιμοποίησε την, περίπου την ίδια διατύπωση, το ίδιο μήκο κύματο. Ωστόσο τα κράτη πρέπει να ενεργήσουν νομίμως και αυτό είναι ένα αγαπημένο θέμα στις εξετάσεις ε, που βάζουν ε, οι καθηγητές σε διεθνούς δικαίου στους φοιτητές τους. Αν δηλαδή αν γίνει μια σφαγή, τα κράτη, τα κράτη μπορούν να παρέμβουν με τη βία. Η απάντηση είναι προφανώς όχι, εκτός και αν ρητός δώσει την άδεια το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, ε, καθηγητά David. Και τώρα το λόγο θα δώσω στον κύριο Σάιμον Άνταμς, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής του Παγκοσμίου Κέντρου για ε, την ευθύνη ε, προστασίας. Ε, το κέντρο παρακολουθεί την εφαρμογή του, της ευθύνης προστασίας. Ευχαριστώ πολύ ε, τόσο τους προέδρους όσο και ε, ε, τους συνομιλητές μας, καθώς επίσης και τα μέλη των επιτροπών που, που βρίσκονται σήμερα εδώ. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πιο ανθρώπινη ιστορία, διότι πολλές φορές ε, όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, πολύ συχνά ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους. Πέρσι το Δεκέμβρη λοιπόν ε, μου ζητήθηκε ε, να εμφανιστώ στο Αλτζαζίρα και να μιλήσω για την πτώση του Χαλιπίου ε, και όπως έκανα και πολλές ε, φορές τα τελευταία πέντε χρόνια έβγαλα το κινητό για να στείλω ένα μήνυμα σε συναδέλφους που βρίσκονται εκεί πέρα για να μου πούν τι πληροφορίες έχουν και τότε συνειδητοποίησα ότι κυριολεκτικά κάθε άνθρωπος που γνώριζα στην πόλη ήταν εκτοπισμένος, είχε εξαφανιστεί, ήταν νεκρός ε, και ήταν μια στιγμή που με έκανε να πάψω ένας από τους συναδέλφους μου είπε ότι ήταν σκοτεινές εποχές. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Προσφύγων και ε, όπως αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή υπάρχουν 65 εκατομμύρια άνθρωποι, άνθρωποι στον πλανήτη που είναι εκτοπισμένοι, ο μεγαλύτερος αριθμός από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και βλέποντας την παγκόσμια κατάσταση συνειδητοποιούμε ότι ε, η παγκόσμια νομοθεσία για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται υπό ε, επίθεση βλέποντας τη δολοφονία αμάχων αλλά και τους βομβαρδισμούς νοσοκομείων όλο αυτό γίνεται καθημερινότητα σήμερα πάνω από το 80% της, ε, των ε, πόρων για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια χρησιμοποιούνται για, τις, για την προστασία από συνέπειες που έχουν προσκληθεί από τους ανθρώπους. Βλέπουμε το Ιράκ, το Νότιο Σουδάν, όλα αυτά επηρεάζουν την ανθρώπια κοινότητα όπως οι πόλεμοι στην πρώην Γιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 90 και ιστορικά κανένα θέμα ε, δεν έβλαψε περισσότερο τη φήμη των Ηνωμένων Εθνών παρά τον, ε, την αποτυχία να σταματήσει ε, τις ε, ε βιοπραγίες αυτές από τη Ρουάντα μέχρι τη Γιουγκοσλαβία. Όλα αυτά λοιπόν υποβιβάζουν τις ιδρυτικές αρχές του ΟΗΕ και θα ήθελα να πω ότι κάποιες χώρες εδώ πέρα, η μεγαλύτερη ζώνη ειρήνης στον πλανήτη, οι φωνές ξενοφοβίας ρίχνουν το να κάνουν αποδιοπομπαίους τράγους ε, τους ε, ε, πρόσφυγες. Όλες αυτές οι φωνές αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και ας μην ξεχνάμε ότι η λέξη γενοκτονία έπρεπε να εφευρεθεί για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους τρόμους οι οποίοι είχαν προκληθεί εις βάρος της εβραϊκής κοινότητας της Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν από μερικά χρόνια στην Στρεβρένιτσα είχαμε άλλη μια γενοκτονία στην Ευρώπη οπότε καταλαβαίνουμε ότι καμία Ήπειρος δεν έχει ανοσία ε, σε αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας ε, προειδοποιεί, να μας ενημερώνει ε, και να καθορίζει τις πράξεις μας. Η ευθύνη προστασίας υιοθετήθηκε το 2005 στη Σύνοδο στην Παγκόσμια Σύνοδο Καρεφής και καταλάβαμε τότε τα μέτρα και τις μεθόδους που υποβιβάζουν, που προκαλούν τις τους μαζικούς τάφους, τις μαζικές δολοφονίες και τώρα έχουμε μια παγκόσμια αποδοχή ε, της έννοιας ότι όλες, ε, όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν τους πληθυσμούς τους από τις εθνοκαθάρσεις, ε, τα εγκλήματα πολέμου, τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Λιβύη και η Συρία αποτελούν τα νεκροταφεία της ευθύνη προστασίας. Όπως αναφέρθηκε από προηγούμενους ομιλητές, τα πέντε χρόνια πριν από το 2001 και την παρέμβαση στη Λιβύη η ευθύνη Προστασία είχε αναφερθεί μονάχα σε τέσσερι αποφάσει του, ε, της Γενικής Συνέλευση του ΙΕ. Έκτοτε όμω έχουν περάσει 42 ε, ε, που αναφέρονται στην ευθύνη Προστασία. και αρκετέ εξ αυτών ε, πέρασαν αποφάσεις για να αποφευχθούν τέτοια θέματα όπως είναι στο Μάλι, στο Σουδάν και η ευθύνη Προστασία λοιπόν έχει επηρεάσει πολύ τι ζωέ ε, ανθρώπων που ζουν στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία αλλά και στην ακτή ε, Ελεφαντοστού. Ε, και οι συνέπειες της Λιβύης μας δίδαξαν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να φυλάτουμε την ε, κακομεταχείριση αρχών. Όμως η πραγματική πρόκληση για την ανθρώπινη κοινότητα είναι ότι θα πρέπει να προστατεύει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και ηρωνικά το ε, βάθος και η ένταση των ε, σειράξεων έχουν καταστήσει την ευθύνη προστασίας ακόμα πιο σημαντική. Υπάρχουν τρεις τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούμε και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερος. Πρώτον, αφορά το ζήτημα της πρόληψης. Η πρόληψη βρίσκεται λοιπόν στην καρδιά της ευθύνης προστασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, εξάλληψη της παγκόσμιας φτώχειας. Χρησιμοποιώντας το στόχο 16 των ε, βιώσιμων στόχων της χιλιετίας θα πρέπει ε, να περιορίσουμε ε, τις σειράξεις όπου ε, οι πολιτικές ταυτότητες, οι ε, μάχες σχετικά με τους πόρους επηρεάζουν τις ευάλωτες κοινωνίες. Βλέποντας τη Μιανμάρ και τον Μπουρούντι μπορούμε να δούμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να μετατρέψουμε την έγκυρη προειδοποίηση σε πρόληψη. Όμως η ανάπτυξη των παγκόσμιων δομών για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών έχουν ε, βοηθήσει ιδιαίτερω. Έχουμε το Σύμβουλο Ειρήνη ε, στην Κάνα, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, όμω και από τη δική μα οπτική, 59 χώρε που απαρτίζουν το 1 τέταρτο των μελών ε, του ΟΗΕ έχουν ορίσει έναν, ένα μέλος της, έναν υπεύθυνο για την ευθύνη προστασίας το Περού, η Καμπότζη, η Ρουμανία, η Νότιο Αφρική, το Τίμορ Λέστερ το Ανατολικό Τιμόρ ε, αλλά και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έναν υπεύθυνο για την ευθύνη προστασίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη η οποία έγινε μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου ε, είδα ότι ο Κρίστιαν μπήκε μόλις τώρα την σωστή στιγμή για αυτό το ε, σχόλιο. Ε, απομένουν πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ορίσουν έναν υπεύθυνο για την ευθύνη προστασία, όμως θα ήθελα να τονίσω και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τον περσινό Ιούνιο 184 ευρωβουλευτές ε, σχημάτισαν ε, το ε, δίκτυο ευρωβουλευτών για την πρόληψη της γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και το δίκτυο αυτό είναι αφιερωμένο για να διασφαλίσει ότι η ευθύνη προστασία εφαρμόζεται και θα ήθελα να τους χαιρετήσω για την αποτελεσματικότητά τους. Πιστεύω ότι περισσότερα μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να γίνουν μέλη αυτής της ομάδας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει οθετήσει επίσης αποφάσεις όπου, οι οποίες αφορούν διάφορα κράτη-μέλη όπου γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η Σύρια, το Ιράν, η Εμένη, οι Φιλιππίνες, το Σουδάν, ε, το ε, Μπουρούντι, η Σομαλία. Αυτό λοιπόν αποτελεί απόδειξη όπως αναφέρθηκε ότι, ότι οι ευρωβουλευτές ε, είναι ανήσυχοι πολίτες ενός μεγάλου κόσμου και η ευθύνη προστασία θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως για παράδειγμα την απόφαση σχετικά με την κατάσταση στην Δημοκρατία του Κογκό ε, και θα ήθελα να γνωρίσω την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η υπηρεσία θα πρέπει ε, να επεμβαίνει σε συνθήκες που αφορούν διαμάχες αλλά και να βοηθά στην ανοικοδόμηση της ειρήνης. Ε, θα ε, πρέπει να υπάρχουν πολυμερείς ε, επαφές διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αποτελεί ο μεγαλύτερος δωρητής προς, τον, προς τις προσπάθειες αυτές του ΟΗΕ και επίσης η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αλλά και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, ενέκριναν ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την αποτροπή γενοκτονιών και την ευθύνη προστασίας. Όταν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να βελτιώσουμε την εικονότητά μας, να ανταποκριθούμε άμεσα. Ο δεύτερος τομέας λοιπόν αφορά την ε, διασφάλιση της ειρήνης. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στις 16 αποστολές του ΟΗΕ που περιλαμβάνουν το 95% των 100 ε, ε, αποστολών. Ε, η προστασία της ειρήνης λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο και σε πάρα πολλές χώρες του πλανήτη αυτή τη στιγμή ε, οι ε, κυανόκρανοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προσπαθώντας να διαφυλάξουν τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Όμως ε, από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι την αποστολή μπορεί να περάσουν μήνες όπου συνεχίζονται να γίνονται τέτοιες αποτρόπες πράξεις. Για παράδειγμα χρειάστηκε ένας χρόνος στον Μπουρούντι μέχρι να φτάσουν στη χώρα. Ε, Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι ε, η αρχή για την προστασία των αμάχων που σχετίζεται άμεσα με την ευθύνη προστασίας και ε, συμμετέχουν χώρες που αποστέλνουν τεύματα. 40 χώρες έχουν υπογράψει αυτές τις αρχές που εκπροσωπούν πάνω από το μισό των αποστολών του ΟΗΕ. Η η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός χρηματοδότης ε, στις αποστολές του ΟΗΕ, όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι σύμφωνα με τους τελευταίους αριθμούς κανένα κράτος μέλος δεν βρίσκεται ε, στο, ε, στα top 20 των κρατών που συνεισφέρουν σε στρατεύματα. Υπάρχουν 7 κράτη-μέλη που βρίσκονται στο top 50 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκήσει πολιτική πίεση στα κράτη-μέλη για να τηρήσουν την ευθύνη τους ε, ως προς την ευθύνη προστασίας. Για παράδειγμα στις 4 Φεβρουαρίου πέρσι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια ομόφωνη απόφαση ούτως σχετικά με, τις, με τα εγκλήματα του ISIS τα οποία θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως γενοκτονία. Επίσης η απόφαση αυτή κάλεσε τα κράτη-μέλη να παράσχουν προστασία και βοήθεια συμπεριλαμβανομένη και στρατιωτικής προστασία σε περιοχές που δέχονται επίθεση από το ISIS. Και πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό ότι αυτοί οι οποίοι ε, διαπράττουν τέτοια εγκλήματα θα αντιμετωπίσουν την παγκόσμια δικαιοσύνη. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με 4 ε, αποστολές όπου συμμετέχουν ε, στρατιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουν στη δημιουργία δυνατοτήτων σε χώρες όπου είχαν γίνει τέτοια εγκλήματα. Και ο τελευταίος τομέας αφορά την ανοικοδόμηση και την τιμωρησία όλα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ε, της όλης προσπάθειας και σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μεγαλύτερο κοινοβούλιο στον πλανήτη το οποίο αναγνωρίζει ε, την ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος ε, και θα πρέπει να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση μετά τη σύραξη και αυτό μπορεί να βοηθήσει ιδιαιτέρως. Μία άλλη ιστορική πρόκληση αποτελεί ε, η ε, μάχη κατά της ατιμορρησίας ε, Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η δικαιοσύνη είναι κολλητική και μπορεί να βοηθήσει στο να τιμωρηθούν οι υπέτειοι θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί όπως ε, στην Αργεντινή και στην ε, Καμπότζη, ε, στη Σενεγάλη που σχετίζονται με αποφάσεις των, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να ερευνήσουν τις, τα εγκλήματα στη Συρία αλλά και να εφαρμοστεί η παγκόσμια νομοθεσία και, όλα, και θα πρέπει να καλέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε και αυτό ε, να, ούτως και στην περίπτωση του Ιράκ να δημιουργηθεί μια τέτοια επιτροπή για να εξετάσει ε, τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται από την πλευρά του ISIS ε, ε, όσον αφορά τον πληθυσμό των γεζίδιδων. Ε, ένα μήνυμα το οποίο πήρα στις 24 Σεπτεμβρίου πέρσι από ένα φίλο μου του Καλίντ στο Χαλέπι μου είχε πει ότι ήταν η χειρότερη μέρα από τις επιθέσεις ε, της ε, Συρίας και την Ρωσία. Μου είπε η το Χαλέπι πεθαίνει, εάν συνεχίσουν οι επιθέσεις όπως σήμερα όλοι μας θα πεθάνουμε, σας παρακαλούμε βοηθήστε μα. Οι άνθρωποι είναι σημαντικοί και τα κοινοβούλια και οι θυσμοί είναι σημαντική και οι ιδέα στο ίδιο. Ζούμε σε δύσκολες εποχές όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάχη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κανόνων που έχουν αναπτυχθεί τον τελευταίο αιώνα για να συνεχίσουν να έχουν σημασία για τους πιο ευάλωτους του πλανήτη. Από τη Συρία μέχρι το Σουδάνι, από τη ε, μέχρι οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, όλα αυτά ε, είναι πολύ σημαντικά. Ο λόγος λοιπόν που εισήχθη η ευθύνη προστασίας δεν είναι επειδή ε, ο πλανήτης ήρθε ένα, μια νέα έννοια. Ήταν εξαιτία τη Ρουάντα, τη Σερβρένιτσα, του Νταρφούρ. Η ευθύνη προστασία προέκυψε επειδή η παγκόσμια κοινότητα αντιμετώπιζε ξανά και ξανά την πραγματικότητα αυτή ε, και σήμερα πάλι η παγκόσμια κοινότητα θα κριθεί από την ικανότητά της να ανταποκριθεί. Έχουμε αποτύχει ανθρώπους όπως είναι ο Καλύψης στη Συρία. Όμως έχουμε μια υποχρέωση να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή της ευθύνης προστασίας στο Κογκό, στο Νότιο Σουδάν, τη Μιανμάρ, αλλά και σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι πάντοτε να ενισχύσουμε αυτό τον σύνδεσμο μεταξύ των ανθρώπων, των ιδεών και της δράσης και πιστεύω ότι αυτό το κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί 700 ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους ε, θα γίνει ένα εργαλείο ε, όπου ιδέες, άνθρωποι και θεσμοί δεσμεύονται ώστε να τηρήσουν την συνολική μας ευθύνη προστασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα έτσι, για την παθιασμένη σας παρέμβαση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις σας που μας θυμήσατε και υπογραμμίσατε ότι αυτό που χρειάζεται πάντα είναι η αναφορά στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες ε, απομακρυνόμαστε από αυτό. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λέφλε, καλώς ήρθατε, ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο και στα μέλη της Επιτροπής μας Έχουμε λίγο χρόνο. Ο κύριος Μπούχνερ, λέω, έχει στήσει το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην τελευταία ομιλία. Για μένα πρόκειται για ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των αποφάσεων του ΟΗΕ ε, και την πρακτική εφαρμογή. Ε, πρόκειται για μια σειρά διαδικασιών που δεν τηρούνται. Θα ήθελα να αναφερθώ στη Γάζα, το, τη Δυτική Ορδανία και πολλά άλλα παραδείγματα τα οποία δεν θα αναφέρω τώρα. Πώς είναι για παράδειγμα παράδειγμα στις κουρδικές περιοχές όπου υπάρχουν πόλεις με άμαχους που βομβαρδίζονται ε, και που πυροβολούνται στους δρόμους ενώ περπατάνε. Δεν ε, έχουμε καμία αντίδραση. Θα είναι, είναι αναγκαίο λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα και πρακτικά να επέμβουμε. Εδώ λοιπόν ο ΙΕ θα πρέπει να αντιδράσει. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Θα μπορούσαμε ίσως να συλλέξουμε καταρχήν όλες τις ερωτήσεις. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως πολλοί που ενδιαφέρονται για ανθρώπινα δικαιώματα, για το σεβασμό τους, την αποτελεσματική εφαρμογή τους, εγώ πάντα πίστευω ότι το ζήτημα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ίσως να είναι και ένα θεμελιώδες ζήτημα, όμως ε, η εφαρμογή, η πρακτική εφαρμογή ε, είναι κάπως ανησυχητική. Η εξέλιξη δεν είναι καλή. Είχαμε κάποια στιγμή κάποιες ελπίδες, όμως σε γενικές γραμμές ε, τα πράγματα δεν τελείωσαν καλά. Και βεβαίως με τη χρήση του άρθρου 7 της χάρτας. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν, να σας ρωτήσω, εν για να μπορέσει αυτό το δικαίωμα, αυτά τα δικαιώματα να εφαρμοστούν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να γίνει. Υπάρχουν νομικά στοιχεία αλλά και πολιτικά στοιχεία. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από αδιέξοδα. Πώς μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και πώς νομικά μπορούμε να προχωρήσουμε και εν τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρα από τα ψηφίσματά μας ε, τα ωραία ψηφίσματα αυτά εγώ προσπαθώ να συνεισφέρω αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει πολλές αρμοδιότητες τους ή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής έχουμε λοιπόν αυτό το όριο ότι κάνουμε απλά ωραία ψηφίσματα τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτό Ευχαριστώ ο κύριος Κρτζίμπ έχει τον λόγο παρακαλώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας σε αυτήν την συνεδρίαση. Έχω ένα ερώτημα για κάποια πρόσφατα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη Συρία, το Ιράκ στα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία, στο Λίβανο. Δείτε παραδείγματο χάρη την Τουρκία. Εάν ισχύουν οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μας, το κύμα προσφύγων έλαβε χώρα σε μια στιγμή όπου η κατάσταση πλέον στα στρατόπεδα ε, των προσφύγων ήταν ανυπόφοροι γιατί δεν υπήρχαν επαρκείς πόροι. Είχαν μειωθεί στο μισό η καθημερινή διατροφή και αυτό οδήγησε στο ότι οι άνθρωποι έρχονται να φεύγουν. Αποφάσισαν να να, να σώσουν τον εαυτό τους, τους κοντινούς τους ανθρώπους και αποφάσισαν να διασχίσουν τη θάλασσα. Πολλοί από αυτούς πέθαναν στην προσπάθεια αυτή. Στα θέατρα επιχειρήσεων επίσης έχουμε δει ε, την ε, ε σφαγή μειονοτήτων οι Γιαζίδοι, οι χριστιανοί στην Συρία, στο Ιράκ, μας περιέγραψαν δραματικά γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πολάκης έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που θα πρέπει να καταγραφούν ως τέτοια και να υπάρξει λογοδοσία σε επίπεδο διεθνού δικαίου. Σε ποιο βαθμό αυτή η ευθύνη προστασίας αντιβαίνει την πραγματικότητα στα στρατόπεδα προσφύγων στην Τουρκία. Υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο. Ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος, όπου δηλαδή υπάρχει η παρέμβαση μιας άλλης χώρας, αλλά δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής αυτής της χώρας. Πώς μπορούμε να ορίσουμε ποιο, τους, τον υπεύθυνο, τους υπεύθυνους σε επίπεδο δικαίου, διότι στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπισμένοι που έχουν φύγει από την περιοχή του Ντόνιετς και του Λουγκάνσκ. Ποια είναι η προσέγγισή σας σε ό,τι αφορά τη θέσπιση αρμοδιότητας. Ναι, παρακαλώ σου γίνεται πιο σύντομα. Ο κύριος Τόκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις στην ακρόαση αυτή. Είδαμε στη Συρία, στο Ιράκ, ότι όταν υπάρχει κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, τα διεθνή φόρα είναι ανίκανα να κάνουν το οτιδήποτε. Και αυτό συνέβη και στη Στρεμπρέντσα Μετά βέβαια έγιναν κριτικές, ε, είχαμε ε, μετάνοιες. Εγώ είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη μνήμη και θα θέλαμε να ε, κάνουμε μία έρευνα για τα εγκλήματα των κομμουνιστών. Όπως την Ιρεβέργη. Στην Ιρεβέργη λογοθότησαν οι Ναζί για τον κομμουνισμό, όμως δεν συνέβη αυτό. Και εδώ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λάβαμε επακή υποστήριξη. Παρότι το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μία απόφαση να, να ληφθεί δράση με σε νομικό επίπεδο. Η ευθύνη προστασίας είναι εξαιρετικά σημαντική αρχή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να το προασπίσουμε και να κάνουμε σοβαρές προσπάθειες σοβαρά βήματα έτσι ώστε αυτή η ευθύνη προστασίας να θωρακιστεί. Σας ευχαριστούμε πάντως για το έργο σας και τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ τον κύριο Τόκες και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Λίφλετ να κάνει την παρουσίασή του. Ε, νομίζω ότι οι ερωτήσεις σας αφορούσαν όλους, μπορείτε να απαντήσετε στο τέλος του τελικό γύρο παρεμβάσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγγνώμη που άργησα. Ήμουν σε μια άλλη διάσκεψη όπου έκανα μια παρουσίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα παρόλα αυτά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Είναι εδώ καλός μου φίλος, ο κ. ο Σάιμον Άνταμς, ο καθηγητής Νταβίδ, αλλά και άλλοι εδώ, τα άλλα μέλη του πάνελ. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε. Επίση, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έχω τη δυνατότητα να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα τη ε, ευθύνη προστασία Είναι κάτι που το κάνω ε, και στα πλαίσια τη περιουσία δράση, δράσης, αλλά, και ω ε, σημείο επαφή ευρωπαϊκό για την ευθύνη προστασία. Είναι κάτι που υπάρχει εδώ. Υπάρχει από το 2016 αυτή η θέση είναι μια πρόκληση για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή ε, με υποφελή τρόπο για τις συγκεκριμένες αρχές και σε επίπεδο των Εθνών. Αναστήσαμε διάφορους τρόπους ε, για να ενσωματώσουμε την εθνική προστασία και την πρόληψη ε, των εγκλημάτων στα πλαίσια της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μέρος των προτεραιοτήτων μας στα Ηνωμένα Έθνη. Το είπαμε και το λέμε κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση από το 2005. Η μεγάλη πρόκληση βέβαια είναι πώς αυτό θα μεταφραστεί σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ακούσατε κάποια πράγματα σήμερα, αποτυπώνονται και αποτυπώνεται και σε ερωτήσεις άλλωστε η απορία αυτή. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους που θα φανούν βεβαίως γραφειοκρατικοί αλλά Είμαστε μια γραφειοκρατία. Έτσι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να εφαρμόσει τις πολιτικές της. Πρώτον, αναπτύσσουμε, ενισχύουμε και προσπαθούμε να διαδώσουμε την πολιτική αυτή δέσμευση σε ό,τι φορά την ευθύνη προστασίας, σε ό,τι φορά την ε, ευθύνη ε, πρόληψης από εγκλήματα. Στη δική μας εξωτερική δράση προσπαθούμε να το ε, αφαρμόσουμε αυτό και προσπαθούμε επίση να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση, την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων. Για το θέμα της πολιτικής βούλησης. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο ε, στις εργασίες μας. Δηλαδή η ύπατη εκπρόσωπος προσπαθεί να το κάνει αυτό ε, στις διαμεσολαβήσεις, στην πρόληψη σειράξεων, προσπαθεί να ε, καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς τις ευθύνες τους και να τις αντιληφθούν. Τώρα, όταν έχει ξεκινήσει μια συλλεξία, όταν τα πράγματα είναι πλέον εκτός ελέγχου, όταν η κρίση είναι στο απόγειό της, πρέπει να μπορούμε ε, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και τα κράτη-μέλη, να τους επιστούμε την προσοχή για να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά, ανθρωπιστικά. Βεβαίως, ε, όταν έχουμε φτάσει πια σε αυτή τη φάση, όπως έχουμε δει δυστυχώς ε, σε, στο, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη, Ορισμένε φορές είναι πολύ αργά. Είναι πολύ δύσκολο να αποτρέψουμε τα εγκλήματα. Η πρόληψη λοιπόν και η πιο αποτελεσματική εργασία νωρίτερα είναι αυτή που μετράει. Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε ένα σύστημα έγκης προειδοποίησης ό,τι αφορά τις σειράξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, να μπορούμε δηλαδή ε, να ερμηνεύουμε μηνύματα ε, και να μπορούμε να αντιδρούμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Είναι όλο και πιο σημαντικό αυτό στις επιχειρήσεις μας επιτόπου Προσπαθούμε δηλαδή να ενσωματώσουμε ενεργά αυτή τη διάσταση της προστασίας των ε, πολιτών και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι τοπικές ε, και εθνικές αρχές ασφαλείας ε, είτε μιλάμε για αστυνομία, είτε μιλάμε για στρατό ότι γνωρίζουν και ότι έχουν εκπαιδευτεί για να μπορούν να λάβουν τις ευθύνες τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λογοδοσία, τέθηκε αυτό το ερώτημα, ε, τι μπορούμε να κάνουμε σε διεθνές επίπεδο γι' αυτό. Πέρα από την κρίση, πέρα από τη σύραξη, υπάρχει το θέμα της ανοικοδόμησης της κοινωνίας και της συμφιλίωσης που είναι απαραίτητη μετά από μια τέτοια κρίση. Θέλουμε να τονίσουμε όμως εδώ την έννοια αυτή της λογοδοσίας. Δηλαδή για να το πούμε απλά, πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη και πρέπει αυτό να φανεί. Πρέπει να γίνει γνωστό για να μπορέσει να υπάρξει εκ νέου εμπιστοσύνη από τους ε, πληθυσμούς. Αυτό παίρνει χρόνο. Μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο. Είδαμε περιπτώσει πρόσφατα στην Αμερική, στην Αργεντινή, στη Χιλή, στην Κεντρική Αμερική, όπου μετά από 30, μετά από 50 χρόνια η δικαιοσύνη φτάνει στους ενόχους. Νόμιζαν ότι ήταν ε, ασφαλής. Αλλά αυτή η ευθύνη δεν χάνεται ποτέ. Παραμένει σύμφωνα με το εθνές δικαίωμα η λογοδοσία και είναι κάτι που έχω συζητήσει συχνά ε, με τους συναδέλφους αφορά ε, αφορά αυτούς που έχουν διαπράξει τα κλίματα αφορά και αυτούς που δεν μπορούσαν να προστατεύσουν γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας είναι λοιπόν μια συλλογική ευθύνη κυρίως αφορά εκείνους στην κοινωνία που δεν ανέλαβαν τι ευθύνε του να προστατεύσουν μια κοινωνία. Αφορά το σύνολο τη διεθνού κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε μια σειρά από επιμέρους εστιασμένες δράσεις οι οποίες μπορεί να έχουν αποτέλεσμα πιο μακροπρόθεσμα όμως. Να δούμε ε, την κρίση στη Συρία. Υπάρχει η Επιτροπή Διεθνή Δικαιοσύνη και Λογοδοσία που συλλέγει στοιχεία ε, και συνεισφέρουμε ε, για τη δημιουργία του νέου μηχανισμού λογοδοσίας της Συρίας ε, έναν ανεξάρτητο μερόληπτο μηχανισμό για να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά θα διαφυλαχθούν εν ώψη του μέλλοντος. Θα είδατε σε κάποια πρόσφατα έγγραφα ότι Αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στις πολιτικές μας, στο προστάσιο μας αν θέλετε. Η ευθύνη προστασίας, η πρόληψη εγκλημάτων πλέον αποτελούν μέρος της ε, παγκόσμιας στρατηγικής που παρουσίασε είπατε και πρόσωπος πριν από λίγο καιρό. Πρόσφατα μια ανακοίνωση για τη δημιουργία αντοχής ε, στις κοινωνίες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορων μορφών σειράξεις ε, και εκεί αναφέρεται η πρόληψη των εγκλημάτων αλλά και στη νέα συνένεση για την ανάπτυξη δίνεται έμφαση σε αυτή τη διάσταση ε, ασφάλεια, σταθερότητα και πρόληψη αποτελούν πλέον μέρος των δράσεών μας και συνεργαζόμαστε με τους συντέρους μας στα Ηνωμένα για να δούμε πώς μπορούμε αυτό σε επιχειρησιακό επίπεδο να το μεταφράσουμε. Το κάνουμε και πολύ συγκεκριμένα αυτό, αναπτύσσοντας ε, μια εργαλειοθήκη που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέλη, ε, τα κράτη-μέλη, οι συνάδελφοί μας, ε, να μπορούμε να εντοπίσουμε τα ευαίσθητα σημεία, τις αδυναμίες και να δούμε από εκεί πέρα τι μπορούμε να κάνουμε, ποια πολιτικά εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά και να μεταφράσουμε τη γνώση που έχουμε σε συγκεκριμένη δράση για δράσεις πρόληψης ε, στα διάφορα πλαίσια όπου μπορεί να εμφανιστεί κάτι τέτοιο. Λίγα λόγια ακόμα για τα ερωτήματα που τέθηκαν. η απογοήτευση ε, που έχει υπάρξει το γεγονός ότι τα τελευταία 10, 12, 15 χρόνια δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά αυτή η έννοια της ε, ευθύνης προστασίας. Ξέρουμε ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολλές στιγμές ε, απογοήτευσης. Όμως δημιουργώντας, ε, οικοδομώντας ένα νέο πεδίο γνώσης, ε, μαθαίνοντας νέους τρόπους να συνεργαστούμε, να συνδυάζουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και θα επανέλθω στο, και επανέρχομαι στο της λογοδοσίας, ε, καθιστώντας σαφές ανά τον κόσμο ότι και οι δράστες αλλά και οι απλοί παρατηρητές θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους ή για τις παραλήψεις τους. Και αυτό δεν παραγράφεται ποτέ με βάση το διεθνές δίκαιο. Ό,τι και να προσπαθήσετε να κάνετε σε επίπεδο μεταβατικής δικαιοσύνης. Και είχαμε κάποια επιτυχία ε, εδώ και δεν έχει αναφερθεί επαρκώς. Θα αναφερθώ μόνο σε μία, επειδή δεν υπάρχει χρόνος. Η διαδικασία ερήνευσης στην Κολομβία. Η Κολομβία έχει ψηφίσει το κείμενο της Ρώμης ο πρόεδρος Σάντο είπε ευθύ εξ αρχή διαδικασία ειρήνευση ότι θα υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία μόνο εφόσον αυτή θα είναι συμβατή με το ICC. Και πολλές φορές ήρθαν εκπρόσωποι τη Κολομβίας, είδαν το ICC, είδαν ότι όλο υπάρχει συμβατότητα με τις διατάξεις περί ε, μεταβατικής δικαιοσύνης στα πλαίσια του κειμένου της Ρώμης. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς το κείμενο αυτό. Αν δεν έχει μετρηθεί με κάποια ευαισθητοποίηση για την ευθύνη προστασίας. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια θετικά στοιχεία. Και κάτι τελευταίο. Έγινε μια αναφορά στην κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία και στο Λίβανο. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να ωρεοποιήσω το οτιδήποτε, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η Τουρκία, ο Λίβανος ή η Ορδανία έχουν αναλάβει τεράστια ευθύνη προσπαθώντας να προσφέρουν προστασία σε ανθρώπους που έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους στη Συρία. Είναι τεράστια η επιβάρυνση και είναι κάτι που πρέπει να το σεβόμαστε. Και με το και το οποίο αξίζει τη συνεργασία μας. Τώρα κάποια στιγμή υπήρξε μια ξαφνική αύξηση το 2015. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε το γιατί. Μπορεί να υπήρξε το θέμα τη διατροφή, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αν δείτε τις εξελίξεις ε, τη ε, σύραξη. Ε, είχαμε και κάποια σημαντικά, σημαντικές εξελίξεις, σημαντικά γεγονότα, η συμμετοχή και κάποιων εξωτερικών παραγόντων άλλαξαν την προοπτική στα πλαίσια ε, της ε, και αυτό μάλλον είχε ε, περισσότερη, περισσότερες επιπτώσεις. Αυτό είναι άλλο επίπεδο ευθύνης προστασίας. Είναι αυτοί που δεν έλαβαν την προστασία που δικαιούταν στις χώρες τους, στις κοινωνίες τους, στις κοινότητές τους. Και εμείς, η Ευρώπη, η Τουρκία, η Ορδανία, ο Λίβανος, και άλλοι οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε και νομικά υποχρεωμένοι από το Σύμβαση της Γενέβης. Είμαστε και ηθικά υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε και να τους υποστηρίξουμε. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει να οδηγήσουμε την κεντρική ευθύνη αυτών που οδήγησαν τους τρόπους αυτούς ε, μακριά από τα σπίτια τους. Ευχαριστώ. Oh, Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ίσως για το τελευταίο γύρο. Εάν μπορείτε να απαντήσετε στα ερωτήματα που ετέθησαν, τρία λεπτά, ο έκαστος, ο κ. Σιμόνοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προσπαθήσω να μοδοποιήσω τα ερωτήματα. Θα έλεγα ότι στην ουσία αφορούν το θέμα της αντίδρασης στις ε, ε, σημερινές προσκλήσεις ανάλογα με την περίπτωση κάθε χώρας και πώς μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η ευθύνη αυτή για την προστασία. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου έχουμε βαθιές αντιπαραθέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτός ο διχασμός ενισχύεται από εθνικά συμφέροντα των μελών και κυρίως των μονίμων μελών. Δεν υπάρχει καμία χρυσή ε, μαγική λύση για το πώς θα λυθεί το θέμα, αλλά μπορεί να ασχεθεί πίεση. Αυτή η ιδέα του να γίνεται ετήσια συζήτηση περί του, περί συγγνώμη, λογοδοσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με την πρόληψη ε, ε, σφαγών γενοκτονιών. Αυτό εκθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας, ε, το κάνει υπεύθυνο, ε, λογοδοτεί και στα άλλα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν το καθένα τις δικές τους υποχρεώσεις και πρέπει να ασκούν κάποιες λειτουργίες. Εάν δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να τους το θυμίσουμε όπως επίσης η ευθύνη για προστασία γεννήθηκε μέσα από τις τραγωδίες της Ρεμπρένιτσα και της Ρουάντα. Η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να κατευθύνεται από τις τραγωδίες της Λιβύης και της Συρίας επίσης. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν λογοδοσία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις δράσεις του, αλλά και για την αδράνειά του. Ανεφέρθη το θέμα ε, ως προς το τι μπορούν να κάνουν οι βουλευτές. Οι βουλευτέ είναι παντού ένα σημαντικός μηχανισμός λογοδοσία που θυμίζει τις κυβερνήσεις τις υποχρεώσει τους και μέσα στο σύστημα του ΟΙΕ θυμίζει Τη Ένωση, μάλλον, σε θυμίζει και στου άλλου θεσμού τι οφείλουν να κάνουν. Και γι' αυτό χαίρομαι για αυτή την παράγραφο που θα περιληφθεί στο δικό σα ψήφισμα και που συστήνει στο Συμβούλιο τι θα πρέπει να αντιπροσωπεύει και τι θα πρέπει να στηρίξει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να σας θυμίζω το ψήφισμα του 2013 και το μακρύ κατάλογο μέτρων που ε, τότε είχατε υπόψη σας. Ορισμένα εξ αυτών έχουν εφαρμοστεί και βλέπω και μια ζωντανή απόδειξη δίπλα μου. Αλλά πρέπει ακόμα κάποια μέτρα να εφαρμοστούν και όπως μου είπαν και νωρίτερα μπορεί να θελήσετε να θεσπίσετε μια ετήσια συζήτηση για αυτό το θέμα ή να χρησιμοποιήσετε τρέχοντα θέματα που συζητάτε στην ημερήσια διάταξη για να δείξετε το θέμα της αξιολόγησης καθώς και της κινητοποίησης των ίδιων πόρων. Είναι καλό που ο Σάιμον μας θύμισε ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα για τους πρόσφυγες και είναι σημαντικό να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στην πρόληψη των εισαγών και την μεταναστευτική ή προσφυγική ροή πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα όσον αφορά τη χορήγηση πόρων το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ και να σας πω ότι ήμουν ευτυχής που άκουσα ε, που θέλετε να μοιραστώ μαζί σας αυτή την παρουσίαση πράγμα που σημαίνει για μένα ότι μπορεί να δοθεί κάποια συνέχεια. Ναι, μπορείτε να είστε βέβαιος ότι θα δοθεί συνέχεια. Όλοι σας κάνατε πολύ λεπτομερείς συστάσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε Καθηγητά Νταβίντ, ε, αν μπορείτε να είστε σύντομος. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε, για να είμαι σύντομος εδώ. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα της αποτελεσματικότητας του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα μεγάλα ε, προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Το κεφάλαιο 7 του χάρτη επιτρέπει πολλά να γίνουν. Ωστόσο, πρέπει να καταφέρουμε να πείσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα μέλη του. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αν σκεφτούμε την τραγωδία της Ρουάντα, ήταν εξαιρετικά εύκολο να ενεργήσει. Αλλά έγινε μια έκτακτη παρέτηση ορισμένων κρατών, μάλιστα και του Βελγίου μέσα σε αυτά τα κράτη, που μάλιστα είχε, είχε πιέσει τον ΟΗΕ να αποσυρθεί από τη Ρουάντα. Ήταν το σκάνδαλο των σκανδάλων. Το Βέλγιο είχε μια μοναδική ευκαιρία να στεφθεί με δόξα και στεφθεί με ντροπή. Αλλά δεν ήταν η μόνη χώρα, γιατί τελικά το σύνολο των χωρών είπαν άστος, άστος να βγάλουν τα μάτια τους μόνοι τους. Τελικά αυτό κάνανε. Ελάχιστα αρκούν. Όχι πάντα για να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά τουλάχιστον να δημιουργηθούν κάποιες ζώνες ασφάλειας. Τα... Σκεφτείτε εκείνο το, με το ξενοδοχείο. 450 όλοι και όλοι είχαν μείνει εκεί. Μόνο και μόνο το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάλαβε, ε, μπόρεσε να διώξει τους ε, δολοφόνους που έρχονταν κάθε μέρα. Απλά τους είπαν δεν μπαίνετε στο δικό μας ξενοδοχείο και σώσαν έτσι 2.000 ανθρώπους. Εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε τώρα πίσω στο παρελθόν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκομίσουμε διδάγματα. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και όντω η διπλωματία των διαδρόμων, ναι, έχουμε πυρογνώμονε εδώ που γνωρίζουν ότι στο καφενείο του ΟΗΕ κάποιε φορέ καταφέρνουμε να κινήσουμε τα πράγματα και είναι μοχλοί που κινητοποιούν, πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε και κάποιε φορέ πετυχαίνουν ε, αυτέ οι προσπάθειε. Ευχαριστώ καθηγητά Ντάιβιτ και τώρα ο δόκτωρο Άνταμ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ που μας ε, κάνατε να αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου με αυτόν τον ωραίο αυστραλέζικο και νοτιοαφρικανικό καιρό που έχει σήμερα έξω. Η Ρουάντα αναφέρθηκε εδώ και εγώ Είχα αυτό το, την αμφίβολη τιμή να δουλέψω στη Ρουάντα μετά από τη γενοκτονία και κάτι που επανειλημμένα ακούγεται από τους επιβιώσαντες της γενοκτονίας είναι το γιατί, γιατί επιτρέψατε να γίνει αυτό και έχουν την αίσθηση ότι επιτράπηκε να γίνει γιατί η Ρουάνδα ήταν κάπου μακριά χαμένη. Ήταν, είναι μια μικρή χώρα, δεν είχε πετρέλαιο και δεν ενδιαφέρονταν κανεί. Να συγκρίνω και την κατάσταση δύο, δεκα, αργότερα σε μια χώρα ε, όπω η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε με τους πρέσβεις ε, του ΟΗΕ για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία δεν ήξερε κανεί που έπεφτε αυτή η χώρα. Ε, μόνο, και μόνο το όνομα τη χώρα του έλεγε ότι είναι κάπου στην Αφρική. Αλλά και πάλι ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας να κινηθεί για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πολύ αργή κίνηση. Ε, οι 10.000 ε, ε, είναι η ειρηνευτική δύναμη εκεί και πάλι μετά με τα χίλια ζόρια. Πάντως όταν τα δεν είναι μόνο όταν πάνε στραβά τα πράγματα που πρέπει να ενεργήσουμε. Η έγκυρη προειδοποίηση, η πρόληψη είναι σημαντική. Και τέτοιε συζητήσει όπω εδώ στο Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικέ γιατί το να μιλάμε για αυτά τα πράγματα έχει σημασία. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να λύσει να προλάβει εμφύλιο πόλεμο, μπορεί να βοηθήσει με τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται η Ευρώπη με αυτό τους, που, τους πρόσφυγες και τους ζητούντες άσυλο, τους άσυλο και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μπορεί να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα για τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και να κλείσω ίσως με μια παρατήρηση που έκανα και στο τέλος της πρώτης μου ομιλίας γιατί νομίζω αυτή είναι η ουσία που θέλω να υπογραμμίσω, ότι πιστεύω πολύ στα ιδέες, στους θεσμούς και στους ανθρώπους, τα άτομα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές. Η φωνή σας έχει μεγάλη αξία. Εμείς σας ακούμε όταν ε, ε, υψώνετε τη φωνή σας και ειδοποιείτε εγκαίρως για το τι μπορεί να συμβεί σε ορισμένες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Ντέιβιντ, τον καθηγητή Άνταμς και τον κύριο Σίμονιτς Ίσως όντως μπορούμε να υιοθετήσουμε κάποια από τα λόγια σας στην εκτίμηση κινδύνου και την πρόληψη. Καμιά χώρα δεν είναι απολύτως ε, ε, προστατευμένη από ε, σφαγές και γενοκτονίες. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Είπατε ότι από τα χαρτιά πρέπει να περάσουμε στη δράση και ορισμένοι είπατε ότι ακούτε, ακούγεται όταν ψώνουν τη φωνή τους οι ευρωβουλευτές. Εγώ δεν είμαι πολύ <laughs> βεβαία γι' αυτό, αλλά ας το ελπίζουμε και ας ε, πούμε ότι είναι έτσι. Είναι δύσκολη καιρή, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και γνωρίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την Συρία, για την Ιεμένη, και να έχουμε υπόψη μας ότι 22 χρόνια πριν μόλις έγινε η σφαγή της Σεμπρένιτσα και το θυμόμαστε όλοι. Πρέπει, πρέπει να δράσουμε. Αυτό είναι ο ρόλος μας των πολιτικών. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε σήμερα και σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και θα κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση των όσων υπόθηκαν σήμερα. Ευχαριστώ και